Παρακαλώ, ο κύριος Σαλάτου. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα η Πρόεδρος Κρόπερκ να είχε παρέμβει και σε παρόμοιες ε, περιπτώσεις για να έχουν απελευθερωθεί και πολιτικό κρατημόνιο στο Ιράκ, πέρα από αυτό που είπε σήμερα.